Καλώς ήρθατε λοιπόν στην επανάληψη της συνεδριάσεως. Τα πρακτικά της χρησινής συνεδριάσεως καθώς και τα εγκεκριμένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Έχετε σχόλια. Δεν βλέπω κανένα να επιθυμεί να σχολιάσει, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη για θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου είναι με πρώτο υποθέμα το Ιράκ και ειδικότερα η θανατική ποινή περιλαμβανομένη στις περιπτώσεις του Ταρί Καζίζ, καθώς και οι επιθέσεις κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, με πρώτο συντάκτη τον κύριο Μπέλντερ, που λαμβάνει το λόγο για 3,5 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Μία εφημερίδα γερμανική πρόσφατα έλεγε διωγμή θανάτου κατά χριστιανών και έδειχνε μια φωτογραφία μιας χριστιανικής οικογένειας που είχε καταφύγει σε έναν ναό στην Βαγδάτη διότι οι Ισλαμιστές τρομοκράτες είχαν αρχίσει να επιτίθενται κατά των οικειών, κατά των σπιτιών ε, χριστιανών. Υπήρξε μάλιστα επίθεση κατά Χριστιανικής Εκκλησίας στις 12 Οκτωβρίου και δεν πρόκειται για μεμονωμένε περιπτώσεις. Οι χριστιανικές κοινότητες ε, στην χώρα των δύο ποταμών, στη Μεσοποταμία, υφίστανται διωγμού. Είναι πραγματικότητα, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Εξού και η ε, μαζική φυγή των χριστιανών. Από το 2003 οι αριθμοί τους έχουν κατέβει από πάνω από 800.000 σε 350 και πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είναι πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Ασφαλώς όσοι παραμένουν εκεί αναμένουν από την Ευρώπη βοήθεια διότι οι χριστιανικές κοινότητες στο Ιράκ χρονολογούνται από τον πρώτο αιώνα με πολλές εκκλησίες, πολλές μονές και γι' αυτό εγώ απευθύνω έκκληση για να υποστηριχθούν οι χριστιανικές κοινότητες που ορισμένοι από τους ε, ανθρώπους αυτούς έχουν καταφύγει στις κουρδικές περιοχές, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται ένα εξασφαλισμένο μέλλον στην χώρα τους. Χρειάζονται βοήθεια και ε, για την ασφάλειά τους και για την επαγγελματική τους εκπαίδευση, χρειάζονται πιστώσεις για να δοθούν σε νέους επιχειρηματίες. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να πιέσουν την Ιρακινή κυβέρνηση να μην ε, εμφανίζει το θρήσκευμα στις ταυτότητες που δίνει στους ε, πολίτες διότι αυτό τους καθιστά αυτομάτως αντικείμενα διωγμού. Οδηγεί λοιπόν σε σοβαρότερες διακρίσεις σε βάρος τους. Τρίτο, τώρα, στο κοινοβουλευτικό επίπεδο θα ήθελα να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της αντιπροσωπείας για σχέσεις με το Ιράκ να τονιστεί το θέμα αυτό, ιδίω σε καιρού αβεβαιότητα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδου κοινοβουλευτικέ επαφέ που έχουμε με το Ιράκ για να ενισχύσουμε την ε, νεαρά αυτή δημοκρατία και χαίρομαι που ο κύριος Μάουρο πρόκειται να ε, υποβάλει έκθεση για το Ιράκ και αυτό είναι σημαντικό. Εν τέλει, απευθυνόμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω, καλά το Συμβούλιο είναι απόν, αλλά τουλάχιστον η Επιτροπή ας καταβάλει προσπάθεια Α έρθει σε επαφή ξανά και ξανά με τις Ιρακινές αρχές ώστε να προστατεύσουν τις χριστιανικές κοινότητες στην χώρα τους. Η κυρία Ντεκάιζερ, 4,5 λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, μετά από τον πόλεμο του Ιράκ, αυτή η χώρα αντί να απολευθερωθεί από μια στρατιωτική δικτατορία βυθίζεται στη βία. Το θέαμα του απαγχωνισμού του Σαντάμ Χουσέιν δεν αποτέλεσε αντικείμενο άμβλησης της βίας, αλλά όξινε τα πράγματα. Ξε, γνωρίζετε ότι είναι αδιάκοπη η μάχη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της θανατικής ποινής. Έχοντας καταργήσει τη θανατική ποινή στην Ευρώπη θεωρούμε ότι συμβάλαμε στο προχώρημα της πρόοδου της ανθρωπότητας. Γι' αυτό λοιπόν η ιδέα της εκτέλεσης διαπαντχονισμού του Ταρέκ Αζίζε και δύο βοηθών του θεωρούμε ότι είναι αποτρόπη όχι λόγω της προσωπικότητας του Ταρικαζής που είναι μια αξιόλογη προσωπικότητα η οποία μπλέχτηκε σε ένα απολυταρχικό σύστημα. Εγώ το γνώρισα προσωπικά και πιστεύω ότι την τελευταία στιγμή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες ε, για να ανοίξει τη χώρα του. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα του Ταρικαζής και να θεωρείται ο απαγχωνισμός του σύμβολο της απολευθέρωσης του Ιράκ. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τους συναδέλφους να υπερψηφίσετε αυτό το ψήφισμα το οποίο σε ένα κομμάτι του αναφέρεται και στις επιθέσεις κατά των χριστιανικών κοινοτήτων στο Ιράκ. Για ένα λεπτό η κυρία το Ιράκ έχει ε, επανειλημμένα παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά αναφέρονται στην ε, Χάρτα των Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων και ε, στη Χάρτα Θημεριδών Δικαιωμάτων. Πάντως, το 2009 18 χώρες αποφάσισαν να καταργήσουν την θανατική ποινή. Το Ιράν, στο Ιράν μάλλον, 388 ε, ήταν οι εφαρμογές θανατικής ποινής ε, και βεβαίως χώρες όπως η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες σε μία τέρμανη λίστα έχουν συνεχίσει να εκτελούν. Ε, οι εκτελέσεις γίνονται στο όνομα της δικαιοσύνης. Όμως καμία σχέση δεν έχει θανατική ποινή με τη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά δεσμευμένη στην κατάργηση της θανατική ποινή οπουδήποτε αυτή ισχύει και προσπαθεί ε, να επιτύχει παγκόσμια αποδοχή αυτής της αρχής. Αποφάσεις ε, σαν αυτή που έχουμε μπροστά μας ε, μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ε, κατάργηση της θανατικής ποινής. Ευχαριστώ. Βαντάλεν για ένα λεπτό. Donkere wolken van moslim-extremisme trekken over de gehele wereld ο εξτρεμισμός με όλες τις φαίες περιοχές του δυστυχώς υπάρχει ακόμα σε πολλές χώρες του κόσμου και στις αραβικές ε, χώρες ακόμα περισσότερο. Ε, οι χριστιανοί δυστυχώς στις αραβικές χώρες και στο Ιράκ συγκεκριμένα ε, είναι αντικείμενο διαρθρωμένων και προγραμματισμένων βίαιων πράξεων και αναγκάζονται σιγά σιγά να εγκαταλείψουν χώρες τις οποίες είχαν εγκατασταθεί πολύ πριν τις καταλάβουν αναλάβουν αυτοί οι εξτρεμιστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεωρήσει την κατάσταση εξαιρετικά επίγουσα. Θα πρέπει να βοηθήσει τις μετριοπαθείς ομάδες στο Ιράκ έτσι ώστε να ενισχύσει την παρουσία της και μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να κλείσει ο κύκλος της βίας των μουσουλμάνων και δεν θα καταφέρουν αυτοί να κλείσουν τις εκκλησίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η ομάδα των πράσινων ΕΦΑ υποστηρίζει το ψήφισμα για την καταδίκη, για την καταδίκη των εκτελέσεων, των θανατικών εκτελέσεων και ζητούμε και εμείς να μην εκτελεστεί η θανατική καταδίκη του Ταρέκα Ζής και δύο συνεργατών του. Ο, πρέπει να καταδικάζονται τέτοιες βαριές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εμείς είμαστε στρατευμένοι σε αυτόν τον σκοπό. Θέλουμε όμως και άλλα πράγματα που δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο. Φαίνεται πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφεύγει να θέσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για περιπτώσεις όπου φέρουμε ευθύνη, διότι τα διεθνή στρατεύματα που βρίσκονται εκεί έχουν κατ' επανάληψη παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη καταδικάστηκε η Μεγάλη Βρετανία από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και η ε, εταιρεία Wikileaks έχει διοχετεύσει δημοσιότητα έγγραφα που ε, μαρτυρούν περί ε, βασανιστήριων και από πλευράς Αμερικανών στρατιωτών. Και έχουν ακουστεί καταγγελίες και για παράνομες απαγωγές και κρατήσεις σε Ιρακινές φυλακές. Οι εξελίξεις που σημειώνονται τελευταία στην ε, Μεγάλη Βρετανία ε, πρέπει να συνεχιστούν, πρέπει ε, να υπάρξουν διώξεις για τα αδικήματα αυτά. Ένα λεπτό, κύριος Πόρτας. Πρόεδρε, Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο να πούμε ότι με αυτήν την απόπειρα εκτέλεσης του Ταρίκαζης ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μια τραγική φάρσα διότι ήδη έχει καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά. Σε αυτό όλοι συμφωνούμε αλλά δεν μπορούμε εμείς να καταδικάζουμε αυτήν την απειλή εκτέλεσης χωρίς να αναφερόμαστε στις πάνω από 900 εκτελές, θανατικές ε, ε, ποινές που εκτελέστηκαν από το Συμβούλιο, το Ερακινό Συμβούλιο, δηλαδή την αρκινή κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά και για τους γνωστούς αλλά και για τους αγνώστους εμείς συμφωνούμε να καταδικάσουμε την Ισλαμική τρομοκρατία κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Αλλά δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε και 30.000 αθώους κρατούμενους στο Ιράκ λόγω της στρατιωτικής κατοχής που δημιούργησε εμφύλιο πόλεμο στην Ιρακινή κοινωνία. Αυτό είναι ένα ψήφισμα που δεν έχει νόημα και γι' αυτό λοιπόν το, η ομάδα μας υποστηρίζει το δικό της ψήφισμα. Η κυρία Λεγκρίπα. θα ήθελα κατά τη συζήτηση για το Ιράκ, την καταδίκη σε θάνατο του Ταρή Καζίκης και την διώξη, τις διώξεις των χριστιανικών κοινοτήτων να εκφράσω την πεποίθηση του ΕΛΚ κατά της θανατικής ποινής. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω όμως και τον αποτροπιασμό μας για την τραγική υποβάθμιση της κατάστασης των χριστιανών στο Ιράκ. Να εκφράσω τη συγκίνησή μας για τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των χριστιανικών επιθέσεων στο Ιράκ, όπως επίσης και την άνανδρη κράτηση ομήρων με 58 ε, θύματα στον καθεδρικό ε, να, ε, καθολικό ναό του Ιράκ. Θα θέλαμε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατευθούν οι χριστιανοί στο Ιράκ, να προστατευθούν όλοι οι τόποι, οι θρησκευτικοί τόποι συνάθρησης όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων και κοινοτήτων και να εργαστούμε προς την ε, μείωση των διεθνικών βίων πράξεων. Πρέπει να προστατεύσουμε τις αρχές της ελευθερίας και της ανοχής. Περνάμε τώρα στου ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Μάουρο από το ΕΛΚ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η θανατική καταδίκη του Ταρίκα Καζίζ και οι συστηματικές διώξεις ε, των χριστιανών στη χώρα αυτή ε, είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά είναι καλό που τα συζητάμε τα δύο θέματα αυτά γιατί θέλουμε να καταδείξουμε ότι θέλουμε ε, πρώτα δικαιοσύνη μέσα στο Ιράκ και δικαιοσύνη για το Ιράκ. Θέλουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα δικαιοσύνη μέσα στο Ιράκ έτσι ώστε να απαγκιστρώσουμε ε, από την ομοιρία στην οποία έχουν περιέλθει από τους Ισλαμιστές φονταμενταλιστές ε, οι ε, χριστιανοί που ζουν στη χώρα αυτή. Θέλουμε επίσης δημοκρατία για το Ιράκ γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την θανατική καταδίκη ενός ανθρώπου που φυσικά ενδεχομένως είναι ένοχος αλλά Όλα αυτά δεν αξίζει να του αφαιρεθεί η ζωή. Νομίζουμε ότι εάν καταφέρουμε ε, να ε, ε, μπορέσουμε να βάλουμε τα θέματα αυτά στο περιεχόμενο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιράκ θα γίνει κατανοητό ότι εμείς θέτουμε προϋποθέσεις και όρους στις εμπορικές συμφωνίες με το Ιράκ. Προϋποθέσεις που αφορούν την, το τέλος θανατικής καταδίκης και την προστασία των χριστιανών του Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές η κυρία Γκόμες για 1,5 λεπτό e sofreram um cortejo de horrores às mãos do ditador. Οι Ιρακινοί έχουν ε, ε, υποφέρει ήδη στα χέρια του δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν και μετά κατελήφθησαν από ε, ε, μια ξένη δύναμη η οποία θα έπρεπε να δείχνει το δρόμο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όμως τότε ξεκίνησαν άλλες φρικαλαιότητες δεν, ε, ε, ε, εμείς δεχόμαστε την δήλωση του Προέδρου Ταλαμπανή ότι δεν πρόκειται να υπογράψει την εντολή εκτέλεσης του Ταρίκα Ζίζε και αυτό μας χαροποιεί. Πρέπει να δείξουμε ότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δεχόμαστε την θανατική ποινή οπουδήποτε και αν αποφασίζεται και οποτεδήποτε και αν εκτελείται. και δεν αλλάζει η θέση μας ε, μόνο γιατί ο Ταρίκα είναι χριστιανός και βεβαίως ε, όπως και άλλοι συνάδελφοι και εγώ καταδικάζω τις ε, βίες επιθέσεις κατά της κατά των χριστιανών του Ιράκ. Πρόκειται για μια κοινότητα η οποία είναι εγκατεστημένη από πάρα πολύ παλιά στην χώρα αυτή. Απ' την άλλη πλευρά ε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι Σουινίτες, οι Σιήτες, οι Μουσουλμάνοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποφέρει τα περισσότερα δεινά στην χώρα αυτή. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των δικαιωμάτων στην ε, Ιράκ και να συζητήσουμε το θέμα και της ε, πιθανικής ποινής με την Ιρακινή Βουλή. Ε, η κυρία Σάκε τώρα, αλλά να πω ότι παρότι καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να μιλήσετε γιατί μιλάτε από καρδιάς για τα θέματα αυτά, να μην ξεπερνάτε το χρόνο σας. Ευχαριστώ. Στο Ιράκ μετά από την Αμερικανική εισβολή το 2003 αναστάθηκαν οι θανατικές εκτελέσεις αλλά ξανάρχισαν το 2004 και από τότε εκατοντάδες έχουν θανατωθεί. Είναι ωστόσο σημαντικό να υπάρξει ασφάλεια για το θέμα αυτό για το μέλλον της χώρας αυτής. Οι πολιτικοί φέρουν σημαντική ευθύνη για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ. Ασφαλώς το προηγούμενο καθεστώς Σαντάμ συγγνώμη, και τα Ρεκαζής και τα φέρει βαρύτατη ευθύνη. Πρέπει ωστόσο τώρα να οικοδομηθεί συμφιλίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινότητα αξιών και ιδίως σχετικά με την θανατική καταδίκη που έχουμε όλοι ασπαστεί την καταργησή της ενώ υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Κίνα, το Ιράκ και το Ιράν εξακολουθούν να ε, την εκτελούν. Ο Ταλαμπανί δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει την εντολή καταδίκης του Ταρικαζής και χαιρόμαστε για το καλό αυτό μήνυμα. Αλλά αυτό θα πρέπει να βασιστεί σε μια κοινωνία κράτους δικαίου όπου θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να ενισχύσει την Ιρακινή κυβέρνηση σε αυτήν την πορεία. Η σταθερότητα του Ιράκ είναι ακόμα εύθραστη και μπορεί να ε, υπονομευθεί από θανατικές καταδίκες που εκτελούνται από, ένα, από το Ιρακινό κράτος. Η συμμετοχή τους στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα βοηθήσει και θα σταθεροποιήσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, ακολουθεί ο κύριος Κοβάλ που όμως νομίζω ότι είναι απόν άρα θα προχωρήσουμε στην κυρία Δεχζιά εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μου η Γκουε δεν προσυπογράφει το κοινό ψήφισμα όπως επίσης δεν υπογράφει και εκείνο για το Θιβέτ. Την πέμπτη το απόγευμα η Ολομέλεια αρχίζει και γίνεται σουρεαλιστική και λόγω του κενού αλλά και λόγω των θεμάτων που συζητάμε και του τρόπου με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Αρχίζουμε και συζητάμε για μία χώρα ή για ένα θέμα με έναν τρόπο που αντιβαίνει τα διεθνή κείμενα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εμείς ισχυριζόμαστε ότι στο όνομά τους τοποθετούμε τα. Διότι οι Ευρωπαίοι Έχουμε μία δυτική γνώμη και άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουμε να επιβάλλουμε τη δική μας γνώμη στους άλλους. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι συμφωνώ μαζί σας για να ε, αντιταχθώ στην εκτέλεση του Ταρέικαζής και τη θανατική ποινή η οποία φύγει ε, πολλά άτομα στο Ιράκ ακόμη και γυναίκες και παιδιά και θέλω να μιλήσω και για τους αθώους κρατούμενους δηλαδή χωρίς, ε, αυτούς που κρατούνται χωρίς δίκη θέλω να μιλήσω για τις κατεχρήσεις ε, του Ιρακινού στρατού και των ε, δυνάμεων κατοχής, θέλω να μιλήσω για τα παιδιά στρατιώτες. Και σε αυτήν τη διεθνή ημέρα για τη, κατά της βία, για, τη, κατά των γυναικών, θέλω να καταδικάσω και την βία που ασκείται κατά των γυναικών. Θέλω επίσης να μιλήσω και για το στρατόπεδο Ασράφ και όλη τη βία που ασκείται εκεί. Και επίσης θέλω να μιλήσω και για το Θιβέτ. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ. Μη εγγεγραμμένος κύριος Όμπερ Στις 10 Νοεμβρίου κυρία Πρόεδρε, σε επίθεση κατά χριστιανών θα ε, φωνεύτηκαν 10 άνθρωποι πριν από λίγο είχε γίνει επίθεση χριστιανική εκκλησία με 40 νεκρούς. Και το αποτέλεσμα είναι να γίνονται διωγμοί κατά 900 περίπου χιλιάδων χριστιανών στο Ιράκ. Και μάλιστα αυτοί οι διωγμοί επεκτείνονται και σε όλη την Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι μια συνολική τάση η οποία δεν συμβαίνει κάπου στον κόσμο αλλά πολύ κοντά στα σύνορα της Ευρώπης και στην Αίγυπτο και δυστυχώς και στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μέσα πίεσης για να καταπολεμηθεί η τάση αυτή. Για παράδειγμα, στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, ήδη από την ε, ε, τουρκική εισβολή έχουν καταστραφεί πολλές χριστιανικές εκκλησίες και μονές. Και δεν μιλούμε για το Ιράκ, μιλάμε για την Κύπρο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται ένα σύστημα monitoring που να παρακολουθεί διωγμούς κατά χριστιανών παντού και να γίνουν μάλιστα και συγκεκριμένες δράσεις. Δηλαδή να περιληφθούν ρήτρε κατά των διωγμών κατά των χριστιανών σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια όταν διώκονται χριστιανοί. Τώρα, για τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Αζίζ. Και αυτός, όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησης του Σαντάμ, έχουν αξίωση να του συμπεριφερθούν με ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και μάλιστα ειδικά σε μια νεαρά δημοκρατία δεν μπορεί να δεχθεί κανείς τέτοια, τέτοιου είδου μεταχείριση. Και εδώ λοιπόν πρέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλυθεί δράση. Σας ευχαριστώ. Οι μεμονωμένοι ομιλητές τώρα. Πρώτα κυρία Ντελάνγκε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ε, βλέπει με μεγάλη ελευθερία τις θρησκείες αλλά το να ε, εκδηλώσει κανείς την χριστιανική θρησκευτική του πίστη στο Ιράκ απαιτεί και προϋποθέτει μεγάλο θάρρος ε, τον και στην Μοσούλ έχασαν τη ζωή τους δύο αδέρφια αλλά και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε σημαντικές ε, βίαιες επιθέσεις ε, κατά χριστιανικών ε, ομάδων. Υπάρχει μια οργανωμένη στρατηγική από κάποιες ε, ε, οργανώσεις ε, και νομίζω ότι δεν μπορούμε πια να μένουμε με δεμένα τα χέρια. Θα πρέπει οπωσδήποτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε, να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να απευθυνθούμε προς την Ιρακινή κυβέρνηση και να απαιτήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά θα πάω και εγώ προς την κατεύθυνση του συναδέλφου Μάουρο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ε, βάλουμε τον όρο και την προϋπόθεση σε κάθε εμπορική συμφωνία ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ε, ε, χριστιανών στο Ιράκ. Ο κύριος Ρέπο, ευχαριστώ πολύ. Είναι τρομερό το να βλέπει κανείς πως οι αθώοι υποφέρουν λόγω της πίστης τους στο Ιράκ. Οι επιθέσεις κατά των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι καταδικαστές όπου και αν συμβαίνουν. Όλοι έχουν την δυνατότητα, πρέπει να έχουν την ελευθερία άσκησης της θρησκευτικής τους πίστης. Δεν θα πρέπει όμως να εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα χριστιανικό μπλοκ. Όλες οι θρησκευτικές θρησκευτικές ελευθερίες πρέπει να προασπίζονται. Όλες οι θρησκείες πρέπει να είναι ελεύθερος, ελεύθερες διότι αυτό θα μας εγγυθεί και σε μια φιλική επίλυση των προβλημάτων. Θέλουμε το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την Ιρακινή κοινωνία για να μπορέσει να παλέψει κατά της βίας και κατά της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να παλέψουμε κατά της βίας υπέρ των ανθρωπίνων αξιών. Και λάμμα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάνω από 50 χριστιανοί δολοφονήθηκαν στο Ιράκ από εξτρεμιστικές ομάδες μέσα σε ένα μήνα. Είναι ιδιαίτερα βαριές οι ευθύνες της ε, νέας Ιρακινής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την ελευθερία, δημοκρατία και ίσα δικαιώματα στα μέλη όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Μόνο έτσι μπορεί η Βαγδάτη να κερδίσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής όπου υφίστανται διωγμούς πολλές παραδοσιακές χριστιανικές κοινότητες και στην Συρία. Είναι πολύ σημαντικό η κυρία Άστον να θέτει το, πρόβλημα αυτό της ανεξιθρησκείας σε κάθε ευκαιρία στην ε, διεύθυνση της εξωτερικής μας πολιτικής και να περιληφθούν και σχετικές ρήτρε στις συμφωνίες μας. Παρέτσκης, ένα λεπτό. Τα τελευταία χρόνια οι χριστιανικές μειονότητες έχουν υποστεί διωγμούς και βία λόγω των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων με βόμβες με επιθέσεις και αναγκάζονται να φύγουν από το Ιράκ. Καταγγέλλω ως εξτρεμιστικές τις ενέργειες αυτές. Η παρέμβαση εκεί και η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γενικά, οι διαιρέσεις σε, βάρος, σε, ε, σε βάση εθνική θρησκευτική ταυτότητα ή θρησκευτικών πεπιθήσεων αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τις ιρακινέ αρχές. Το ίδιο θα πρέπει οι Ιρακινές αρχές να εγκαταλείψουν την θανατική ποινή. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την δήλωση του Ιρακινού Προέδρου σχετικά με, την, με το δεν θα υπογράψει την εντολή ε, Εκτέλεση του Ταρεκαζή. Ο κύριος Πόσελτ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, μετά από 2.000 χρόνια παρουσίας των χριστιανικών κοινοτήτων στο σημερινό Ιράκ, είναι πραγματικό σκάνδαλο ότι σήμερα και ειδικά μετά από παρέμβαση εκεί του λεγόμενου δυτικού κόσμου, κινδυνεύουν, απειλούνται με εξαφάνιση. Δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Πέραν από τα θέματα, τα γενικότερα θέματα της ανεξιθρησκείας πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι τον Δεκέμβριο θα προσέλθουν εδώ στο Στρασβούργο ένας αριθμός Ιρακινών επισκόπων για να μας ενημερώσουν σχετικά με την κατάσταση των κοινοτήτων τους εκεί. Ας έχουμε σαφώς υπόψη ότι εδώ δεν μπορούμε απλώς κάπου κάπου να κάνουμε μια διακριτική χειρονομία προς το μέρος τους. Είμαστε υπεύθυνοι. 80% των Ευρωπαίων είναι χριστιανοί. Ασφαλώς και τα σώμεθα υπέρ της ανεξιθρησκείας. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών. Άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν ακόμα και του βάρβαρου καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ρίξει ιδιαίτερο βάρος στις προσπάθειές του και απευθύνω έκκληση στην Λέδη Άστον να πράξει το ίδιο και να μας ενημερώνει τακτικά για την κατάσταση των χριστιανών στο Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Αρκετά αιτήματα βάσει τη διαδικασία Catch the Eye. Σόνικ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χριστιανοί δολοφονήθηκαν και δολοφονούνται στο Ιράκ, στην Ινδονησία, στο Σουδάν και ποιος ξέρει που αλλού. Χριστιανοί θύματα βίαιων επιθέσεων που υποχρεούνται πλέον να κρύβουν την πίστη τους. παρότι αυτή η πίστη έχει, είναι βαθιά ριζωμένη και οι άνθρωποι αυτοί είναι ριζωμένοι στις περιοχές τους πολύ περισσότερο από ότι το Ισλάμ. Ο ακρεφνής ε, Ισλαμισμός, οι εξτρεμιστές οδηγούν ε, ολόκληρες κοινότητες ε, σε αφανισμό. Και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν εάν οι μουσουλμάνοι, αν αντιμετωπίζαμε τους μουσουλμάνους σε άλλες χώρες όπως στις μουσουλμανικές χώρες αντιμετωπίζονται οι χριστιανοί. Τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει οπωσδήποτε να συζητώνται στις εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Θεωρώ ότι είναι απολύτως παράλογο να σκοτώσει, να δολοφονήσει κανείς κάποιον μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι δεν είναι καλό να ε, σκοτώνει κανείς. Εμείς ε, είχαμε εξαιρετικά υπηρετική στάση απέναντι στο παλαιό καθεστώς ε, του Ιράκ και βεβαίως βλέπουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν να αλλάξουν τα πράγματα, οι βίες επιθέσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Υπάρχει ακόμα βία και βία κατά των χριστιανών. Αυτό πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ε, ε, ευθύνες του και εμείς απέναντι σε αυτό που ας το ονομάσουμε, ας το με το όνομά του, είναι ε, ξεκαθάρισμα εθνικό θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν είναι δυνατόν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ε, γυρίζουμε, επιστρέφουμε Ιρακινούς στο Ιράκ ενώ ξέρουμε πόσο θα υποφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Οι προθέσεις που κινούν την Ιρακινή κυβέρνηση μπορεί να είναι καλές και θετικές αλλά εμείς θέλουμε να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των χριστιανικών κοινοτήτων που υφίσταται διακρίσεις που μέλη της φωνεύονται υπάρχει και κάποιο όριο. Μιλούμε για μια χώρα όπου οι χριστιανικές κοινότητες έχουν μακρότατη παράδοση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με καθαρή φωνή και όχι αυτολογοκρινόμενη. Σημαίνουν σημαντικές αλλαγές στο Ιράκ και πολλές από αυτές είναι θετικές. Όμως Η κατάσταση αυτή αποτελεί απειλή για την συνέχιση των διπλωματικών σχέσεων της χώρας αυτής. Merci. Οι χριστιανοί είναι ίσως μία από τις, χριστι... μία ομάδες που διώκονται περισσότερο ανά τον κόσμο. Στη Μέση Ανατολή οι ακραίες ομάδες θεωρούν ότι είναι νόμιμοι στόχοι, διότι θέλουν να τους διώξουν από την περιοχή. Περιοχή στην οποία γεννήθηκε ο χριστιανισμός και όπου η ιστορική τους παρουσία είναι απαραίτητη για, για το κράτημα μιας ισορροπίας. Η επιθέση στον καθεδρικό της Βαγδάτης αποτελεί το, το αποκορύφωμα μιας κατάστασης η οποία κρατάει για καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμπορικός και οικονομικός εταίρος πολλών χωρών αυτής της περιοχής και θα πρέπει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε εμείς να ανεχθούμε τις διακρίσεις. Θα πρέπει να νικήσει η δημοκρατία σε αυτές τις περιοχές, αλλά αυτό θα γίνει μόνο όταν θεμελιώδη δικαιώματα όπως η θρησκευτική ελευθερία θα γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να υψωθεί η φωνή αυτού του Κοινοβουλίου για τις επιθέσεις κατά των χριστιανικών επιθέσεων στο Ιράκ. Πρόκειται για μια, ε, διαρκή κατάσταση διακρίσεων και μαρτυρίων που διατηρεί χιλιετίες. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μετριοπαθείς ομάδες του Ιράκ, τους χριστιανούς που έχουν, ε, ε, που, που, που, που κρύβονται ε, πρέπει σίγουρα να, να, να βγάλουμε από τις ταυτότητες την αναφορά για τις θρησκείες. Για τους χριστιανούς το, σύμ, το σύμβολό τους είναι ο σταυρός που δεν είναι σύμβολο θανάτου αλλά είναι σύμβολο ζωής διότι απελευθέρωσε τον, μέσα από την Ανάσταση το Χριστό από την, από, την κόλαση. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να δολοφονούμε κάποιον ο οποίος φέρει το σταυρό και μπαίνει σε μία εκκλησία μόνο για το λόγο ότι είναι χριστιανός. Ο Επίτροπος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σημερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις απόψεις που τόσο καθαρά ε, εξέφρασαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στο Ιράκ. Ήδη το Συμβούλιο της ε, Δευτέρας εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις καλά, κατά συγγνώμη, αμάχων, κατά χριστιανών οι οποίοι βρίσκονται σε ειρηνικές θρησκευτικέ συναθρήσεις και βεβαίως και η ε, Πρόεδρος κυρία ε, Άστον ε, υπογράμμισε την ανάγκη να συζητηθούν ενδελεχώς τα θέματα αυτά και την ανάγκη το Ιράκ να προσυπογράψει το προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνού Συμφώνου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα βασική ε, αρχή θα πρέπει και μεγάλη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία ε, των ατόμων που ανήκουν ε, σε μειοψηφίες. Ε, και βεβαίω όταν μιλάμε για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ δεν αναφερόμαστε μονάχα στην προστασία ε, τη ανεξιθρησκεία αλλά και ε, την κατάργηση τη θανατική ποινή. Έχουμε αντιδράσει στην απόφαση των Ιρακινών δικαστηρίων να στείλουν στην Αγχώνη τον κύριο Ταρίκ Αζής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά ρητά την αντίθεσή της προς ε, την θανατική ποινή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως ε, έχουν σημαίνοντα ε, ρόλο στις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ. Από το 2003 στα πλαίσια της ε, συνεργασίας ε, με το Ιράκ εστιάσαμε την προσοχή μας ε, στις ατομικές ελευθερίες και τις και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω ή λέξε και μέσω συγκεκριμένων πιστώσεων για τον σκοπό αυτό. Ε, μέσω της προσπάθειάς μας έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την, ε, ε, την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε σχολεία και οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναφερθεί ε, σε συγκεκριμένες, στην προστασία συγκεκριμένων ε, μειονοτικών ομάδων αλλά ε, ε, κατανοούμε ότι είμαστε σε θέση να θέσουμε προϋποθέσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα, τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα ε, και θα πρέπει να καταδείξουμε πράγμα που θα κάνουμε στην κυβέρνηση του Ιράκ ότι οι ανεξέλεγκτες δράσεις μεμονωμένων περιθωριακών ομάδων κατά αμάχων δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν γιατί δεν αξίζει στον ε, στο λαό του Ιράκ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση όλης της ε, συζήτησης. Το επόμενο θέμα λοιπόν της σημερινής διάταξης είναι το Θιβέτ. Σχέδια